Eh Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στο σχέδιο προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έτος 2020 και δίνω το λόγο ευθύ αμέσω στον εισηγητή μας, τον κύριο Μάνκα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ήταν απαραίτητο να συμφωνήσουμε όσον αφορά τα νούμερα, τις περικοπές. Χαίρομαι που πετύχαμε συνένεση σε επίπεδο σκιωδών εισηγητών. Μία εκκρεμότητα υπάρχει που εξαρτάται από απόφαση της Επιτροπής μας σχετικά με τις 51 ε, θέσεις που αφορούν ε, τα γραφεία συνδέσμων ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, μπορεί να αναζητήσουμε συμβιβαστικές προτάσεις. Αυτό πρέπει όμως να γίνει κατόπιν συζήτησης. Για παράδειγμα, μπορούμε να διατηρήσουμε έναν συμβασιούχο ανά κράτος μέλος και έτσι να πετύχουμε σημαντικές περικοπές. Μετά από τη συνάντησή μας ε, καταλήξαμε στα εξής. Προ, προτείνουμε περικοπές ύψους σε 18,1 εκατομμυρίων ευρώ με την εκκρεμότητα όσον αφορά τους συμβασιούχους για τα γραφεία συνδέσμου στα διάφορα κρατημέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν συμφωνήσουμε με την περικοπή αυτή, τότε θα έχουμε αύξηση ύψους 2,68% αντί για 3,2%. Υπάρχουν κάποια αιτήματα. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που δεν στηρίζουν την πρόταση της έκθεσης. Θα ήθελα όμως να πω, σε όλους να πω ότι τελικά θα υπερισχύσουν οι, ε, τα ποσοστά που προτείνει η δική μας Επιτροπή, τα χαμηλότερα ποσοστά δηλαδή. Επίσης ε, υπήρξαν διάφορες προτάσεις. Έχουμε τις εκθέσεις Experience Europe, όπου κάποιοι έχουν στηρίξει κάποιες τροπολογίες, άλλοι όχι. Υπήρξαν τροπολογίες στα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούν το θέμα αυτό από μόνο τους, ή αυτό αναζητήσαμε συμβιβασμούς και το συζητάμε με τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Υπάρχει Υπάρχει η απόφαση του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2018, όπου υποστηρίζουμε πρωτοβουλία σχετικά με ε, τις περαιτέρω εξελίξεις μετά το 2019. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις στα διάφορα κράτη-μέλη, ώστε όταν λύγει μία σύμβαση να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σχετικά κτίρια και για τους σκοπούς αυτούς. Υπήρχαν, υπήρξαν όμως διάφορες ε, διορθώσεις ε, και γι' αυτό θα ήθελα από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει την Επιτροπή μας σχετικά με το πού βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να λάβουμε σχετική απόφαση. Για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο άνοιξε ένα κέντρο Experience Europe στο Ελσίνκι ε, και μέσα στον πρώτο 1,5 μήνα λειτουργίας του είχε πάρα πολλούς επισκέπτες ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενημερώσει όσο γίνεται περισσότερους πολίτες σχετικά με το πώς λειτουργεί ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους ανθρώπους να συμμετάσχουν και στις εκλογές. Άλλο σημαντικό θέμα ήταν οι κινητές εγκαταστάσεις για το Experience ε, Europe. Αυτό υποστηρίχθηκε και από το Προεδρείο. Σε κάποια μικρά κράτη-μέλη πιθανότατα να είναι δυνατόν να υπάρξουν μόνο κάποιες τέτοιες κινητές εκθέσεις. Μπορεί για παράδειγμα να έχουμε ένα πούλμαν, να γίνονται επισκέψεις σε σχολεία και να μπορέσουμε έτσι να μεταφέρουμε πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό το υποστήριξε το Προεδρείο, γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή μας να στηρίξει την πρόταση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, υποσχέθηκα να σας ενημερώσω σχετικά με τις διπλωματικές αντιπροσωπίες, κάτι που επίσης υποστηρίχθηκε από το Προεδρείο. Τα μέλη του Προεδρείου στις 14 Ιανουαρίου συζήτησε το θέμα. Όσον αφορά την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ε, σε κάποιες απόμακρες περιοχές θα πρέπει όμως ε, καταρχάς να επικεντρωθούμε σε κάποια ε, συγκεκριμένα μέρη, για παράδειγμα την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά τον αριθμό υπαλλήλων δεν χρειαζόμαστε νέους υπαλλήλους. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στις περιφέρειες όπου ήδη έχουμε αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το, Προεδρο, το Προεδρείο στήριξε την πρόταση να επικεντρωθούμε στις υπάρχουσες επιστολές ΑΣΕΑΝ, Αφρικανική Ένωση και Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. και κατά τη δημιουργία της ε, γνωρίζαμε ότι θα λειτουργεί με υπαλλήλου ε, της Κομισιόν ε, και του Συμβουλίου, αλλά τελικά αποφασίστηκε να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αντιπροσωπείες αυτές. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε νέο προσωπικό, δεν χρειαζόμαστε νέες θέσεις προσωπικού, ούτε νέες εγκαταστάσεις. θα έχουμε κάποια νέα κτίρια στο Λουξεμβούργο. Και υπήρξαν σχετικές τροπολογίες το 2020 να πετύχουμε εξοικονόμηση με μεταφορά κάποιων ε, σε άλλα κτίρια. Αυτό απαιτεί χρόνο και την εξοικονόμηση αυτή θα την πετύχουμε μόλις το 2021. Έχουμε ετοιμάσει όμως συμβαστική πρόταση, όπου ζητάμε από τον Γενικό Γραμματέα να μας υποβάλει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά υπαλλήλων και γιατί δεν είναι δυνατόν οι εξοικονομίες αυτές να επιτευχθούν ήδη το 2020 και αυτή η τροπολογία υποστηρίχθηκε γενικά. Κατόπιν έχουμε το κτίριο PHS. Σε τέλος της χρονιάς θα πρέπει να λάβουμε απόφαση σχετικά με το αν θα το καταργήσουμε ή αν θα το ανακαινήσουμε. Ό,τι απόφαση όμως και να λάβουμε, θα πρέπει να εκενώσουμε το κτίριο και όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να μεταφερθούν αλλού. Έχουμε υποβάλει σχετική τροπολογία. όπου ζητάμε η δική μας Επιτροπή να ενημερωθεί σχετικά με τους υπολογισμούς δαπανών πριν πάει το θέμα στην Ολομέλεια το φθινόπωρο. Αυτή είναι η τροπολογία μας για να λάβουμε συγκεκριμένες πληροφορίες παρότι ήδη έχει ενημερωθεί το Προεδρείο. Άλλο πρόβλημα είναι η προφορική ανακοίνωση των ψηφοφοριών. Άκουσα από διάφορους συναδέρφους ότι πιθανότατα να υποστηρίξουν την κατάργηση αυτών των προφορικών δηλώσεων. Έχουμε ετοιμάσει σχετική τροπολογία και θα πρέπει να εξετάσουμε το κόστος, το οποίο υπολογίζεται σε 800.000 ευρώ το χρόνο. Ζητάμε περαιτέρω τεκμηρίωση και θα αποφασίσουμε εάν είναι κάτι το οποίο τελικά θα καταργηθεί ή όχι. Οι ευρωβουλευτές έχουν εναλλακτικά μέσα στη διάθεσή τους, ε, μπορούν γραπτώς να επεξηγήσουν την ψήφο τους. Πιστεύουμε ότι αυτές οι προφορικές επεξηγήσεις ε, δεν είναι απαραίτητες, αλλά... Αυτό θα εξαρτηθεί από την, από την αποφασή μας. Επίσης, ε, συνταξιοδοτικό ταμείο και στη δική μας επιτροπή συζητήθηκε το θέμα αυτό. Έχουμε εκπονήσει τροπολογία και θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι έχουμε ένα καθεστώς των βουλευτών και η ΑΛΔΕ και το ΕΛΚ έχουν υποβάλει διορθωτικές τροπολογίες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε συμβιβαστική πρόταση ε, που να ακολουθεί το καθεστώς των βουλευτών, όπου λέει ότι το συνταξιοδοτικό ταμείο θα παραμείνει σε λειτουργία και σύμφωνα με το καθεστώς των βουλευτών που υιοθετήθηκε το 2009 και θα υπάρξει εγγύηση των δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν λέει το καθεστώς των βουλευτών και καλούμε το, τη Γενική Γραμματεία να τηρήσει το καθεστώς και να υποβάλει συγκεκριμένα σχέδια για το μέλλον. Επιπλέον, απαιτούμε το ελεγκτικό συνέδριο και στο μέλλον ε, να μας υποβάλει προτάσεις σχετικά με τη διατήρηση του Συνταξιωτικού Ταμείου. Επιπλέον, ε, ε, αγώνας κατά της παρενόχλησης. Έχουμε λάβει πολλά η υπόψη μας ε, στα σχετικά νούμερα που έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε την ιατρική υπηρεσία, χρειαζόμαστε διαμεσολαβητή, ψυχολόγο. Και 161.000 προβλέπουμε να χρειαστούν για εμπειρογνωσία, παροχή συμβουλών κλπ. Έχουμε υποβάλει και εδώ σχετική τροπολογία. Στην έκθεσή μας ζητάμε επίσης ο Γενικός Γραμματέας να επικεντρωθεί στη διοργανική συνεργασία, κάτι το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει σε περαιτέρω εξοικονομήσεις. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε κίνητρα στη διοίκηση για κάτι τέτοιο και να δημιουργήσουμε και σχετικό κλίμα στο Κοινοβούλιο. Εάν μπορούμε να πετύχουμε επιπλέον εξοικονόμηση σε κάποιους τομείς, τότε μπορούν στο τέλος της χρονιάς ε, οι εξοικονομημένοι πόροι να μεταφέρονται, για παράδειγμα, στην κτηριακή πολιτική ή να διατίθενται ε, για συγκεκριμένα έργα του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Δίνουμε έτσι κίνητρο στους υπαλλήλους να πετύχουν εξοικονόμηση μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό θα αποτελεί λοιπόν κέρδος ε, για την κάθε Γενική Διεύθυνση. Αυτά από μένα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιγητά. Για να δούμε οι σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Ρούμπικ ίσως ανέθεσε σε κάποιον άλλον, στον κύριο Φερνάντες, όχι, όχι. Ωραία. Ο κύριος Κόλμπερ τότε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας ε, για την εκτενή εισηγησή του και την πολλή δουλειά που έχει κάνει. Νομίζω ότι έχει παρουσιάσει πολύ σωστά πολλούς ε, τομείς και εάν προβληματιστούμε θα διαπιστώσουμε ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, έχει κάποια αναπόφευκτα στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να τροποποιήσει κανείς, ούτε θα έπρεπε να το κάνει αυτό, εφόσον θέλει να διασφαλίσει τη λειτουργία του. Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, αναφέρθηκαν αυτές, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια. αλλά και όσον αφορά τον σωστό εξοπλισμό, όχι μόνο των Ευρωβουλευτών αλλά και των βοηθών τους, συνολικά του προσωπικού του Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε καλό και ασφαλή εξοπλισμό. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν είχαμε σκάνδαλο για τα δεδομένα. Θα ήταν πολύ η σημαντική η ζημιά σε μια τέτοια περίπτωση, γι' αυτό δεν θα πρέπει να ε, ε, κάνουμε εξοικονομήσεις στον τομέα αυτό. Αντιθέτως, θα πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα αυτό. Προβλήματα όμως έχω όσον αφορά την δημιουργία περαιτέρω θέσεων στο Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι γενικά συμφωνούσαμε στις προηγούμενες ψηφοφορίες ότι πρέπει να έχουμε μία έδρα του Κοινοβουλίου. Άρα δεν είναι λογικό να λέμε ότι πρέπει να έχουμε αντιπροσωπεία σε κάθε κράτος μέλος. Δεν, δεν επιτρέπεται να είναι αυτό ο καθήκον του Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα οι πολιτικές ομάδες, όπως και ο κάθε ευρωβουλευτής που έχει εκλεγεί εδώ, θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά με το Κοινοβούλιο. Ήδη προσφέρουμε πολλές πληροφορίες επιγραμμικά και δεν ε, θεωρώ ότι μπορούμε να δικαιολογήσουμε απέναντι στους πολίτες ε, το άνοιγμα αντιπροσωπιών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό νομίζω θα θεωρηθεί σπατάλη και είναι λάθος μήνυμα να στείλουμε. Σας καλώ να μην κάνουμε κάτι τέτοιο. Merci. Ευχαριστούμε. Ο Ζεράρ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι Σκιώδης. Είμαι απλώς συντονιστής. Αλλά οι επαφές με την κυρία Γιατεμάκη, τον κύριο Μάνκα και λοιπούς, ε, έγιναν μέσα σε πολύ καλό κλίμα. Εγώ θέλω να πω ότι βάση των όσων μου ανακοινώθηκαν και που υπενθύμισε και ο κ. Μάνκα τώρα, συμφωνούμε με το συμβασμό ο αριθμός 8, αν δεν απατώμε, για την όχληση, το harassment, η προσπάθεια που έγινε για τη διατύπωση, αλλά και για το πολιτικά σωστό όσον αφορά το συνταξιδοτικό ταμείο, είναι μια προσέγγιση πολύ καλά ισορροπημένη. Είμαστε ανοιχτοί σε προβληματισμό για την τροποποίηση του συστήματος ε, των ε, αιτιολογήσεων ε, των ψηφοφοριών που μπορεί και να καταργηθούν και κατά τα άλλα όπως εισηγητής έτσι και εμείς τέτοια σκεφτόμαστε. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο έχω κάποιες ερωτήσεις ακόμα γιατί με την ανησυχία που μόλις παρουσίασε και ο κύριος Κόλμελ για τον πολλαπλασιασμό των κέντρων Europa Experience. Ακόμα και αν τροποποιήθηκε το κείμενο σε σχέση με το προηγούμενο που είχαμε. Επί της ουσίας, αυτό που λέει ο συνάδελφος είναι λογικό. Έχουμε όμως εδώ ένα πρόβλημα που είναι, θα έλεγα, θεσμικό ουσιαστικά. Αν έχω σωστές πληροφορίες, πήρα απόφαση το Προεδρείο. Μάλιστα, λέει ότι είναι της 16 Απριλίου του 2018 η απόφαση αυτή του Προεδρείου, που λέει ότι θα υπάρχουν κέντρα Europe Experience σιγά σιγά σε όλες τις χώρες μέλη. Ποια είναι η λειτουργία της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι να πηγαίνει στο Προεδρείο Έτσι, τι ρόλο έχει. Αποφασίζει το Προεδρείο για τα πάντα και για τις δημοσιονομικές συνέπειες των αποφάσεών του ή είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών που έχει αυτή την ευθύνη. Εγώ προσωπικά έχω επιφυλάξεις σε σχέση με αυτόν τον πολλαπλασιασμό των κέντρων αυτών. Και άκουσα τις επεξηγήσεις του κύριου Μάνκα για τη Τζακάρτα και για Λου. Δεν θα υπάρξει επιπλέον προσωπικό. Ναι, αλλά τι θα κάνουν εκεί οι άνθρωποι. Δηλαδή τι, θα στέλνουμε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις ε, πόλεις του κόσμου, σε αυτά τα experience centers. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στρατηγική μας τι είναι η στρατηγική μας επ' αυτού και κανένας δεν μου το έχει εξηγήσει μέχρι τώρα ικανοποιητικά. Μα καταλάβατε ποια είναι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρωτάει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ντεπρέ, κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι πολύ σκληρός, είμαι ήδη λίγο σκληρός. Μα είναι εκπληκτικό, λέει ο Πρόεδρος Αρτουή. Δεν έχουμε αρμοδιότητες. Κάνουμε σαν η Ευρώπη να διακινδυνεύει να δώσει ένα θέαμα ε, για την ε, έλλειψη ικανοτήτων της. Μα εμείς εδώ συζητάμε για τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ για αυτό το πράγμα θέλω να μιλήσω. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω ποια είναι η στρατηγική μα. Θέλω κάποιο να μου την εξηγήσει. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά τη κάνει τα ίδια και το Συμβούλιο από την πλευρά του τα ίδια, με επιπλέον τις 28 πρεσβείες που έχουμε περίπου σε όλες τις χώρες του κόσμου, συν την πρεσβεία της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, εγώ θέλω να καταλάβω, απλώς αυτό θέλω να καταλάβω και δεν καταλαβαίνω. Δεν μου φαίνεται αρκετά σόφρον. Ε, είναι μια απόφαση του Προεδρείου, οπότε εγώ θέλω να ξέρω εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή Προϋπολογισμών για μια απόφαση του ε, Προεδρείου. Αν εμείς δεν επιτρέψουμε τα κονδύλια, τι γίνεται. Αυτά. Ε, τι άλλο. Ε, επέμεινα για την μείωση των κονδυλίων. Ο κύριος Μάκα δεν ξέρω αν είπε το ποσό. Ίσως να ήμουν αφηρημένος εκείνη τη στιγμή. Πάντως πιστεύω πως με τίποτα η αύξηση του προπολογισμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 2,5. 2,5 μονάδες παραπάνω. Με τίποτα. Πρόεδρος, ο κύριος Μάνκα δύσκολα θα τα χωρέσει όλα αυτά και θα μπορέσει να τα συμβιβάσει. Καλώς. Δεν βλέπω άλλο και ο δεσηγητή να ζητάει το λόγο. Οπότε τώρα ποιος θέλει το λόγο. Έχω ότι είναι η καρδιά Μπαζάλ πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Σίγουρα ο κύριος Μάνκα ξέρει πολύ καλά τι κάνει και σίγουρα θα καταφέρει να τετραγωνίσει τον κύκλο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, πάντως δεν είναι η πρώτη φορά και ήταν και δήμαρχος στην περιοχή του, οπότε σίγουρα ξέρει πολύ καλά πώς κάνει κανείς ένα προπολογισμό. Τώρα, εγώ ζήτησα το λόγο πρώτον και μια που μιλάω αμέσως μετά τον κύριο Ντεπρέ, να πω για τη συζήτηση που έχουμε σε όλη αυτή την θητεία. Δηλαδή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αποφάσεις του Προεδρείου που είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές. Απλώς να ε, επιτρέψουμε αρκετά κονδύλια για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Οπότε δεν ξέρω είναι θέμα νομιμότητα, σίγουρα όμως είναι θέμα αρμοδιοτήτων τι αρμοδιότητες έχει το Προεδρείο και τι μπορεί ή δεν μπορεί να αποφασίζει η δικιά μας Επιτροπή. Τώρα, εγώ ζήτησα το λόγο όμως, γιατί έχω ένα σχόλιο και μία ερώτηση όσον αφορά τις 51 θέσεις ε, επικοινωνίας. Το πρώτο μου σχόλιο είναι η εσωτερική επικοινωνία που δεν έχει λειτουργήσει καλά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί όταν εδώ στην Επιτροπή μας μας μίλησαν για τις 51 αυτές θέσεις, όταν πάρθηκε η απόφαση, μας είπαν ότι πρόκειται για ενίσχυση εν ώψη των ευρωεκλογών. Τα ψάξαμε και φαίνεται ότι δεν είναι αυτό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μας εξηγούν από την αρχή ποια είναι η βασική ιδέα. Ότι δηλαδή η επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνει προσπάθειες για να φτάσει πιο κοντά στον πολίτη, άρα στους ψηφοφόρους, κάτι το οποίο προφανώς και είναι αναγκαιότητα. Αλλά μας είχαν πει ότι η προσπάθεια αυτή έπρεπε να γίνει ευθύ αμέσω εν ώψη των ευρωεκλογών, αλλά δεν μας είχαν πει ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιζόταν και μετά. Οπότε κάτι δεν πήγε καλά εδώ στην εσωτερική επικοινωνία. Πρέπει να ξέρουμε πραγματικά ποιος είναι ο στόχος και δεν θα μπω τώρα στο περιεχόμενο ε, του έργου των 51 ε, συμβασιούχου. Προφανώς, μεγαλύτερη παρουσία στα μέσα ενημέρωση, ε, συνεδριάσεις, σεμινάρια, ένα σωρό πράγματα οργάνωσαν, ακριβώς επειδή ενισχύθηκε η υπηρεσία αυτή επικοινωνίας. Και τώρα έρχομαι στις ερωτήσεις μου. Γιατί επιπλέον έχει να κάνει με μία μεταφορά ε, κονδυλίων που θα δούμε μετά με τις προφορίες και με τον προπολογισμό του 2020. Και ελπίζω να έχουμε εδώ και κάποιον από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου για να μου απαντήσει. Λοιπόν, για την μεταφορά 2019 μας ζητούν 3 εκατομμύρια 312.000 ε, για τους ε, μήνες που μας μένουν. Ε, εμένα δεν μου βγαίνει. Δεν ξέρω αν κάτι έχω χάσει για τα 3.312.000 και για το 2020 τώρα. Διατηρούμε αυτήν η πρόταση τους 51 συμβασιούχους και η ε, Διεύθυνση Επικοινωνίας για να αντισταθμίσει ακριβώς αυτήν την ενίσχυση των τοπικών ε, γραφείων θα μειώσει κατά 51 θέσεις τη δίκησή της. Οπότε οι συμβασιούχοι η προσωρινή πρέπει να είναι πιο φτηνή από τους μόνιμους. Έτσι, έτσι υποτίθεται. Οπότε δεν καταλαβαίνω. Αν υπάρξει αυτή η αντιστάθμιση το 2020, τελικά καταλήγουμε σε 4 εκατομμύρια παραπάνω. Δεν ξέρω αν μέσα σε όλο αυτό το σχήμα μου λείπει εμένα κάποια μεταβλητή ή δεν κάνω σωστά τους λογαριασμούς μου. Θα ήθελα πάντως να μου το εξηγήσει κάποιο αυτό. Γιατί νομίζω ότι όλες οι πληροφορίες που έχουμε για την μεταφορά αυτού του κονδυλίου δεν παίζει ρόλο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται για τον ε, προπολογισμό του 2020. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι. Θέλω οι εκπρόσωποι της Κομισιόν να μας δώσουν ε, κάποιες απαντήσεις. Κυρία Ρούμπε, από τη Γενική Διάθεση Κόμμα. Δεν ξέρω πού είναι. Ευχαριστώ. Ο Γενικός Διευθυντής δεν θα μπορέσει να έρθει. Είναι σε αποστολή στην Κοπενχάγη σήμερα. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του. Ε, το Προσαρμόστηκε η απόφαση για την ενίσχυση των γραφείων το 2017. Τα γραφεία λαμβάνουν μια ενισχυμένη εντολή και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερη επαφή με τους πολίτες, τους stakeholders, ε, επαφή με τα ΜΜΕ, τα εθνικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Επομένως, λογικό είναι, λόγω και των εκλογών, η Επιτροπή σας να ζητήσει μια μεταφορά το Φεβρουάριο, ζήτησε μάλλον μια μεταφορά το Φεβρουάριο του 2018, ούτως ώστε να αρχίσει να ε, προσλαμβάνει συμβασιούχους. Ε, τους, αρχίσαμε τους προσλαμβάνουμε τους 51 συμβασιούχους και τώρα κάνουμε την πρώτη αξιολόγηση της δουλειά και είδαμε ότι η Γενική Διεύθυνση Κόμψ ε, έχει μεγαλύτερη επαφή τώρα με τους Δήμους και τις κοινότητες, ε, με τον κόσμο. Υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία κατά 31% σε όλες τις πλατφόρμες, αν συγκρίνουμε το 2017 με το τι γίνεται το 2018 τι έγινε το 2018. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το δίκτυο. Ίσως ε, έχετε έρθει και σε επαφή με το προσωπικό. Στη Μαδρίτη ενισχύσαμε και το γραφείο μας. Ε, θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους κρατήσουμε, ε, τους υπεύθυνους για την επικοινωνία, γιατί βλέπουμε ότι η δουλειά τους έχουν, έχει άμεσο αποτέλεσμα στην επαφή μας με τον κόσμο. Αυτή η μεταφορά που ζητάμε τώρα θα πρέπει να μας επιτρέψει να κρατήσουμε αυτό το προσωπικό για μέχρι το τέλος του 19. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σύμβαση μέχρι τον Ιούλιο. Αρχικά είχαμε τα απαραίτητα κονδύλια για να τους προσλάβουμε μέχρι τις εκλογές. Μέχρι δηλαδή την προεκλογική εκστρατεία και μέχρι να τελειώσει αυτή. 31 ε, Ιουλίου δηλαδή του 2018 και τώρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι κονδύλια για να καλύψουμε τους μήνες από τον προπολογισμό του 20 έχουμε προβλέψει και στον προϋπολογισμό του 20 να κρατήσουμε αυτούς τους συμβασιούχους. Δεν υπάρχει άμεσο ισοδύναμο με τους μόνιμους. Νομίζω ότι αυτή ήταν η ερώτησή σας, δηλαδή να κάνω μια αντιστοιχία με τους, μόνις, με τους μόνιμους. Ε, κάποιοι ESD ε θα αλλάξουν θέση. Ε, γιατί βλέπουμε ότι η δουλειά στα γραφεία αλλάζει και χρειαζόμαστε από, πολύ περισσότερους από αυτού τους ειδικού ε, για θέματα επικοινωνία και τύπου να ασχοληθούν με τον κόσμο, να έχουν επαφή με τον κόσμο και μπορούμε να εξοικονομήσουμε και α, λεφτά που σπαταλάμε στους ASD. Γι αυτό, αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να μετακινήσουμε ASD στα γραφεία. Επίσης, ένας άλλος λόγος που θέλουμε να κρατήσουμε αυτούς τους ε, ειδικευμένους ε, συμβασιούχους είναι ότι αλλάζει η δουλειά των γραφείων και πρέπει να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Κάνουμε αυτή τη μετακίνηση δηλαδή. Από τους ASD στα, στα γραφεία, από, το, από τη θέση που είναι σε, στα γραφεία. Ο κύριος Ντεπχέ. Μία ερώτηση, Πρόεδρε. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα καλά. Και θα ήθελα η Διευθύντρια να με διορθώσει αν δεν κατάλαβα καλά. Μας είπε ότι αυτά τα 51 άτομα δουλεύουν αποτελεσματικά. Γιατί ε, υποτίθεται ότι η επαφή αυξήθηκε κατά το output, ας πούμε, με τον κόσμο δηλαδή, ε, αυξήθηκε κατά 21%. Τι είναι αυτό δηλαδή, μέσω των εκπομπών, είναι Δηλαδή, α, περισσότερα άρθρα για μας. Πώς μπορούμε να το αποτιμήσουμε αυτό, χάρη στη δουλειά, ας πούμε, του, των 51 ανθρώπων. Ε, έγινε κάτι, ας πούμε, με τους Ιταλούς εκλογής, άρχισαν να ανησυχούν, λόγω, ας πούμε, της Τη νέα κυβέρνηση, ε, Ξέρω ότι υπήρξαν προβλήματα στην Πολωνία κτλ. Ε, πώς μετράμε αυτό το output. Είναι θετικά άρθρα ας πούμε, υπέρ τη Ευρωπαϊκής Ένωση στον τύπο ή είναι απλώς μία αύξηση του αριθμού των άρθρων ή εκπομπών που αφιερώνουμε, αφιερώνουν τα ΜΜΕ στην Ευρώπη. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Έχω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις. Δεν είναι απλό ε, να επικοινωνήσουμε υπάρχουν διάφοροι οίκοι Ευρώπης, ας πούμε, έτσι, που έχουν σαν σκοπό να φέρουν σε επαφή τους πολίτες με την Ευρώπη, να τους εξηγήσουν τι έκανε η Ευρώπη. Πρόσφατα, μάλιστα, στη δική μου εκλογική περιφέρεια και μάλιστα στο δικό μου διαμέρισμα στη Γαλλία, ε, ο οίκος για την Ευρώπη οργάνωσε μια συνεδρίαση για να εξηγήσει και να γιορτά... εξηγήσει την Ευρώπη και να γιορτάσει την 20η επέτειο από τη δημιουργία του. Δεν είχε όμω το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει ότι υπήρχε εκεί ένας ευρωβουλευτή. γιατί αυτό ήταν εναντίον της ανεξαρτησίας, ας πούμε, της πολιτικής ανεξαρτησίας υποτίθεται του οίκου αυτού. Εγώ, εντάξει, σέβομαι ας πούμε, αυτή την απόφαση να έχουμε και άλλους ε, υπαλλήλου, για να επικοινωνούμε, αλλά τότε τι γίνεται. Αποκόβουμε, ας πούμε, το πολιτικό στοιχείο, την πολιτική διάσταση από τον κόσμο. Κυρία μου, ποιο είναι το δόγμα σε αυτά τα θέματα, πώς λειτουργεί το πράγμα, τι οδηγίες δίνεται ε, σε αυτούς που παίρνουν τις επιχορηγήσεις, ας πούμε όπως τα οίκη της Ευρώπης για να οργανώνουν ας πούμε, τις δημόσιες ε, εκδηλώσεις τους, τις συνεδριάσεις τους κτλ. Ευχαριστώ. Ίσως να μπορέσω εγώ να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα στον κύριο Ντεπρέ να διαβιβάσω την ανάλυση μας του Δεκεμβρίου του 2018, όπου εξετάσαμε τα αποτελέσματα των σεμιναρίων για δημοσιογράφους που οργανώσαμε, συνεντεύξεις τύπου και ενημερώσεις, briefings. Όσον αφορά τη δημιουργία επαφών, εξετάσαμε την κάλυψη σε, στα μίντια σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή τηλεόραση, κοινωνικά μέσα δικτύωσης, όλα δηλαδή. Και δεν εξετάζουμε αν είναι θετικά ή αρνητικά τα αποτελέσματα, απλά κοιτάμε το σύνολο των επαφών. Όσον αφορά τον οίκο της Ευρώπης, το Maison δεν μπορώ να σας απαντήσω. λαμβάνουν επιχορήγηση, αλλά νομίζω ότι την λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από τη Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν μπορώ να απαντήσω λοιπόν στην ερώτηση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάρας από τη Γενική Διεύθυνση ΦΙΝΣ. Πρόεδρε, Έχετε κάποια ερώτηση για μας? Πρόεδρος, όχι, από αυτά που ακούσατε. Μήπως έχετε κάτι να διευκρινίσετε, δεν θα το θεωρούσατε θεμητό, για να μας εξηγήσετε εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποια είναι η θέση σας. Καλώς, θα σταματήσουμε εδώ γι' αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μάνκα. Δεν ήταν εύκολο το έργο του, σίγουρα. Κύριε Μάνκα, μήπως εσείς θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέρφων. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα απαντήσω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για... Να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά για την παρουσία σας στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Ε, πάντα αποτελεί πλονέκτημα η παρουσία σας, έτσι ήταν και στο παρελθόν. Είναι πολύ πιο αποτελεσματική εργασία όταν είστε παρόν. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Ε, συζητήσαμε σχετικά με τις 51 θέσεις ε, στον τομέα της επικοινωνίας εξοικονομήσει μας ε, δεν έχουν σχέση με το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί ξεχωριστά μετά. Αλλά κάποιες ερωτήσεις δεν απαντήθηκαν. Κάποια γραφεία σε κάποια κράτη-μέλη ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη ανήκουν στις διάφορες χώρες. Στις περιπτώσεις που ανήκουν στο κοινοβούλιο ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο και εξαρτώνται από τον αριθμό των πολιτών στο κάθε κράτος μέλος. Δεν εξετάζουμε όμως κατά πόσο το κτίριο ανήκει σε εμάς ή όχι. Εάν υποστηρίζουμε την πρόσληψη των 51 αυτών ανθρώπων, θα πρέπει να εξετάσουμε ε, αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη ε, και αυτό το θέμα στο μέλλον. Ο κύριος Κόλπελ και ο κύριος Εντεπρέ αναφέρθηκαν σε διάφορες επιτυχίες. Ε, ένα από τα θέματα αυτά ήταν το Experience Europe και τους εκθεσιακούς χώρους. Είπαμε ότι μπορεί να είναι οι διπλωματικές αντιπροσωπείες. Ο κύριος Κόλπελ αναφέρθηκε σε αυτές και θα ήθελα να πω το εξής πραγματικά δεν θα μας στοιχήσουν τίποτα. Έχουμε ήδη υπαλλήλου του Κοινοβουλίου, θα χρειαστούμε χώρους οι οποίοι όμως ήδη βρίσκονται στην κατοχή του Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο υποστήριξε τη δράση αυτή και μιλάμε για περιορισμό αριθμό ε, υπαλλήλων που θα υποστηρίξουν τις εργασίες. Τις δαπάνες που μοιραζόμαστε με άλλα θεσμικά όργανα θα τις εκμεταλλευτούμε με καλύτερο τρόπο με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, Πρόκειται για ένα θέμα συνεργασία δεν θα μας στοιχήσει τίποτα, δεν θα προσλάβουν με νέους ανθρώπους, ούτε χρειαζόμαστε νέες εγκαταστάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τα συγκεκριμένα στοιχεία, συμφωνώ ότι ο προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να αυξηθεί με ποσοστό άνω του 2,8%. Τα στοιχεία που έχουμε εμεί είναι 2,68% και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να περιοριστούμε σε μια τέτοια αύξηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Το θέμα που μας μένει είναι η σχέση αρμοδιότητες μεταξύ Προεδρείου και Επιτροπής Προπολογισμών. Το ερώτημα αυτό θα λήξει θητεία και δεν θα έχει απαντηθεί. Και ίσως θα έπρεπε κάποια μέρα δεδομένων των αρμοδιοτήτων του προεδρίου του Κοινοβουλίου, ίσως να πρέπει μέσα στο Προεδρείο να υπάρχει μια Επιτροπή Προϋπολογισμών και η δικιά μας Επιτροπή ως τέτοια να μην έχει πια αυτές τις αρμοδιότητες, γιατί εφόσον έρχονται και μας λένε «Μα αποφάσισε το Προεδρείο», οπότε μπορώ να φανταστώ ε, πόσο μας ενοχλεί εμάς ε, εδώ όταν είναι το σφυράκι του Προεδρείου που αποφασίζει και εμείς απλώς υπογράφουμε. Υπάρχει μια αμφισημία εδώ. Δεν θα βγούμε από αυτή την αμφισημία όμως στη δικιά μας τη θητεία. Ας το αφήσουμε σαν κληρονομιά στους διαδόχους μας. Ωραία, κύριε Μάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές. Και ευχαριστώ για το κονδύλι που έχει όρια που εξηγούνται. Γιατί όλα τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις χώρες μέλη, εντάξει υπάρχουν, αλλά εμείς πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις να δίνουμε. Ωραία, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα περνάμε στην έκθεση του Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες και του Ρομπέρτο Κουαρτιέλη, που είναι ο συνεισηγητής, έτσι, για το Invest EU. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε ήδη κάνει δύο τριμερείς ε, διαλόγους για το InvestEU. Έχουμε πιέσει το Συμβούλιο, το περιμέναμε πολύ καιρό για να έχουμε εντολή. Στο Συμβούλιο ακόμα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για το πού θα είναι η γραμματεία και θα έχουμε τριμερή διάλογο σήμερα το βράδυ που θεωρώ σημαντικό προβλέπεται και ένα τελικό τριμερής διάλογος για την Τετάρτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί το στόχο του, που είναι να ολοκληρώσουμε το θέμα κατά τη διάρκεια αυτής της θητεία. Το ίδιο είχαμε πει και για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Από τη δικιά μας την πλευρά είμαστε πάντα έτοιμοι, διαθέσιμοι, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία εάν η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η εντολή μας δεν τηρούνται. Από πλευρά του Συμβουλίου πιστεύω ότι επίσης υπάρχει η επιθυμία, η πρόθεση να προχωρήσουν και να ολοκληρωθεί το ζήτημα. Τώρα μένουν θέματα όπως είναι η διακυβέρνηση. Θα σας πω ποια είναι τα πιο δύσκολα. Το θέμα της εγγύησης, το οποίο δεν θα συζητηθεί, γιατί ο στόχος μας αντί για 38 δισεκατομμύρια ε, προτείνονται 40,8 γιατί θέλουμε ακριβώς να διατηρήσουμε την ίδια εγγύηση για τους 14 δημοσιονομικούς ε, μηχανισμούς που τώρα μπαίνουν σε ένα ενιαίο μηχανισμό. Οπότε από αυτού εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάντως το θέμα της εταιρική σχέσης, της συμφωνίας αυτής με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν έχει καταλήξει ακόμα σε συμφωνία. Παραμένουν θέματα σε κρεμότητα. Η δικιά μας θέση είναι να αποφύγουμε σύγκρουση συμφερόντων. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε τέτοια σύγκρουση. Τώρα πώς θα προχωρήσει αυτός ο τριμερής διάλογος, θα δούμε. Αλλά ελπίζω, αν μη τι άλλο, να καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία έτσι όπως προβλέπουμε τουλάχιστον. Τίποτα όμως δεν θα κλείσει αν δεν έχουμε συμφωνήσει επί των πάντων. Με εξαίρεση την εγγύηση, όπως σας είπα πριν. Συμφωνήσαμε σε αυτό πολλές φορές μέχρι τώρα. Πρόεδρο, ωραία. Έτσι καλώς θα είναι προσωρινή συμφωνία, σωστά. Γιατί όσο δεν έχουμε συμφωνήσει για το σύνολο των προγραμμάτων και για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα, σωστά. Βέβαια, αλλά όσο να είναι, αν μπορούμε να προχωρήσουμε και να συμφωνήσουμε μετά αυτό που θα λείπει, ε, ωραία, το, λέει ο Πρόεδρος. Τα οι εισηγητές. Η... Κύριε Καπναζαμάλ. Κολμέλ. Όχι. Κανείς. Ο κύριος Στολβατς δεν είναι εδώ. Σολέ. Όχι. Κύριε κυρία Τριάδα δεν την βλέπω. Ποιος άλλος? Κανείς? Ε, τότε. Χωσέ Μανουέλ καλή επιτυχία σήμερα το βράδυ στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, δεν είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου για το σχέδιο ρύθμισης, για τα μέτρα που θα πρέπει να πάρουμε λόγω του Brexit Οπότε, κάποια άλλη στιγμή θα τα δούμε αυτά. Η ψηφοφορία αναβάλλεται. Δεν έχω να σας πω τίποτα από αυτού προς το παρόν. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει κάποιες ενδείξεις ή όχι. Όχι, ούτε εκείνη. Ένα. Ε, Ίσως όμως θα έπρεπε να προβλέψουμε στον προϋπολογισμό την παρουσία Βρετανών Ευρωβουλευτών από την 1η Ιουλίου και μετά. Ε, μήπως. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Αν βέβαια η Ευρωπαϊκή οπως πάντα τα πραγματα αν αντιστέκεται, θα δούμε. Λοιπόν, ψηφοφορία τώρα. Οπότε βάλτε τις κάρτες σας παρακαλώ στα ηλεκτρονικά μηχανήματα για την ψηφοφορία. Θα κάνουμε πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ωραία, για ψηφίστε. Για τη δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Έχουμε απαρτία. Για να δούμε. Κοιτάξτε. Έληξη ψηφοφορία. Και δίνω το λόγο στον ε, Ντανιέλ Βιώτη, που είναι ο γενικός μας εισηγητής και θα μα παρουσιάσει τέσσερι μεταφορέ κονδυλίων που έχουν να κάνουν με το τμήμα 3 του προπολογισμού του 2019. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, υπάρχουν τέσσερις αιτήσει ε, για μεταφορές ε, από την ε, Κομισιόν. Θέλω να σας πω ότι δύο από αυτές τις αιτήσει έχω πρόβλημα εγώ. Και θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, θέλω να πάω σημείο προς σημείο, μου επιτρέπετε, και να σας παρουσιάσω αυτές τις τέσσερις αιτήσει. Πρώτον, ένα κάθετος 2019. Δεν έχω πρόβλημα. Ε, μεταφορά που αφορά τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την ε, βιώσιμη αλία και το πρωτόκολλο που υπογράφτηκε 14 Ιανουαρίου του 2019 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου για, μέσω της ε, έγκρισης του Συμβουλίου. 37 εκατομμύρια ευρώ θα μεταφορθούν και θα με βάση τη συμφωνία της 10 ης Φεβρουαρίου του 2019. Όπως σας είπα, αυτό το αίτημα δεν, έχει κανένα, δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Ενώ για το υπαριθμό 5 κάθετος 2019, για την αίτηση 5 κάθετος 2009, για τη μεταφορά 5 εκατομμυρίων ε, από το εργαλείο εταιρικής σχέσης στο εργαλείο DCI για την αναπτυξιακή συνεργασία ε, για την ε, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Νοτιού Αφρικής για την διανομή κρασιών και αλκοολούχων ποτών στη Νότια Αφρική με σεβασμό των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω κάποιες ερωτήσεις που θέλω να θέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση την ανάλυση που έκαναν οι συνάδελφοι της ΔΕΒΕ, δεν θεωρείται δεδομένο ότι η στήριξη για τον άμπελο τομέα καλύπτεται από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, το παράρτημα του προγράμματος ε, για το 2018 βλέπουμε ότι ο ε, κλάδος αυτό δεν καλύπτεται από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πρόγραμμα του 2018 αφορά τα δικαιώματα εργασίας, κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη κτλ. κτλ. Θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν Πώς ε, δικαιολογεί ε, ότι αυτά τα 15.000 ευρώ, που είναι ένα ελάχιστο ποσό, από τα 5 εκατομμύρια ευρώ της μεταφοράς θα πρέπει να δοθούν σε μια χώρα σχετικά πλούσια μέσω της ε, στήριξης του προπολογισμού. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα υπόλοιπα ερωτήματα θα τα θέσω μετά. Πολύ ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει στο ερώτημα του κυρίου Βιώτη Κατάλαβα, Πρόεδρε, ότι η συμφωνία για τα 15 εκατομμύρια ήταν τμήμα της ε, συμφωνίας ε, για την εμπορική και αναπτυξιακή συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Νοτιού Αφρικής. Επομένως, με κατέλαβε εξαπίνης ο εισηγητής. Δεν έχω επιπλέον πληροφορίες για να σας δώσω, κύριε εισηγητά, πάρα αυτά. Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες, πρέπει να σας απαντήσω γραπτός τι επόμενε μέρε όχι τώρα. Εν τέτοια περιπτώσει μπορούμε να βάλουμε και την ψηφοφορία. Κύριε Βιώτη, τι λέτε, συμφωνώ. Αναβολή λοιπόν. Πολύ ωραία. Θα μας παρουσιάσετε το σημείο 7. Το 7, το νούμερο 7, ε, θέλει θέλουμε να μεταφέρουμε 1 δισεκατομμύριο 400 εκατομμύρια δεσμεύσεων, ε, πιστώσεων. Όχι, διορθώνει ο μιλητή, όχι ένα, ένα δι. Ένα εκατομμύριο είναι. Για να καλύψουμε τα επιπλέον έξοδα σε ό,τι αφορά την, ε, όσον αφορά το πρόγραμμα Black Book της Κομισιόν για την ε, δυνατότητα να δώσουμε περισσότερες ε, υποτροφίες σε μαθητευόμενους Αυτό ε, λήφθη υπόψη από την πρώτη διορθωτική επιστολή Νομίζω ότι αν μας δώσει μια απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε αυτό το σημείο ακόμα και σήμερα. Μιλάμε για, την, για τα λεφτά αυτά για τους μαθητευόμενους. Έχετε απάντηση η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Βιώτη για την ερώτηση αυτή. Είναι θέμα χρονισμού αυτό κυρίως. Η συμφωνία μεταξύ του Ναύρατσης, του Επιτρόπου Ναύρατσης μάλλον, για την αύξηση βαθμιαία του ποσού για τους μαθητευόμενους ελήφθη αρκετά καθυστερημένα μέσα στη χρονιά, γι' αυτό δεν συμπεριληφθεί την πρόταση. Ε, τα επόμενα, οι επόμενες δόσεις αύξησης για το 2020 όμως θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο προπολογισμού για το 2020. Αν κατάλαβα καλά, ο κύριο Ότιγκερ δεν έδωσε γρήγορα την απάντηση. Τον μια συμφωνία ανάμεσα στου Ναύρατζη και Ότιγκερ. Κανοποιηθήκατε, κύριε Βιώτη. Με το ερώτημά σας, ναι. Va Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. μπορούμε να ψηφίσουμε. Για το 7 δηλαδή θα ψηφίσουμε που δεν υπάρχει πρόβλημα. Για την μεταφορά υπαριθμών 8. Εδώ είχα κάποια ερωτηματικά προς την Επιτροπή για την 8. Θέλω να παρουσιάσω την απόφαση στους συναδέλφους για να μεταφέρουμε 370.000 ε, ευρώ από τις δεσμές πιστο, ε, για να ε, χρηματοδοτήσουμε τον, ε, το άσυλο και τη μετανάστευση στην Ελλάδα. 66,6 εκατομμύρια στην Ιταλία και στην Ισπανία 4 εκατομμύρια. Θα πάνε από το ΑΜΙΦ στο καταπιστευτικό ταμείο Αφρικής 30 εκατομμύρια επίσης. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα στην Κομισιόν για να μου διευκρινίσει καλύτερα την κατάσταση. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε τρεις κατηγορίες, έτσι, θα τα ταξινομήσω. Έχω τρεις διαφορετικές ερωτήσεις. Πρώτον, πώς αποφάσισε η Κομισιόν την κατανομή αυτή των 300, ε, 340 ε, εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ Ιταλίας, Ισπανίας και Ελλάδας. Ε, επιπλέον, ποιες είναι οι αναλογίες μέσω των εθνικών προγραμμάτων άμυ, δηλαδή το, το ΑΜΗΟΥ, Ασύλου και μετανάστευση και πώς η, ε, η Κομισιόν αποφάσισε ποιε είναι οι ανάγκε και ποια είναι η κατανομή των τελικών ποσών. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν, στην κυρία Μπεάτ Κουίντερ, από την DG Home. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εξηγήσω το θέμα αυτό, καθώς και τις πολύ σκόπιμες ερωτήσεις σας σχετικά με αυτό το αίτημα μεταφοράς. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο ε, ε, προγραμματισμό για τις εν λόγω χώρες, χώρες που επηρεάζονται από μεταναστευτικές ροές σε μεγάλο βαθμό και που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών συνόρων λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουμε ένα ε, δημοσιονομικό σχέδιο, το οποίο ε, έχουμε συζητήσει το οποίο συζητάμε με τις ελληνικές αρχές κάθε μήνα, όπου κάποιος ε, ανώτατος υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Home συναντιέται με τις ελληνικές αρχές όσον αφορά το προγραμματισμό, ο οποίος καλύπτει το εθνικό σύστημα του Ταμείου Μετανάστευσης και Ασύλου, διότι γνωρίζετε ότι τα ποσά χωρίζονται στα χρήματα που δίδονται στα κράτη-μέλη σε έναν ετήσιο φάκελο για να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές ε, συν τη δυνατότητα συμπλήρωσης από το ΆΜΙΦ με επίγουσα βοήθεια. Και αυτή έχει πολύ σαφή ορισμό στη νομική πράξη του Ταμείου Ασύλου μπορούν να δοθούν εάν υπάρχει δυσανάλογη πίεση και κάποια επίγουσα κατάσταση. Και όλοι γνωρίζετε από τα στοιχεία ότι πράγματι αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Ουσιαστικά, λοιπόν, προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σε κάθε χώρα, πρώτα μέσω τεχνικού προγράμματος και μόνο όταν διαπιστώσουμε ότι αυτό δεν αρκεί και το εθνικό πρόγραμμα αυτό χωρίζεται σε διάφορους στόχους, προσφεύγουμε σε συμπληρωματική χρηματοδότηση. Η επίγουσα αυτή βοήθεια θα πρέπει να εγκριθεί μετά από μια εντελεχή διαδικασία ε, εξέτασης και ο ετών είναι είτε κάποιο Εθνικό Υπουργείο είτε κάποιος διεθνής οργανισμός. Ε, Πολύ μεγάλο μέρο λοιπόν τη βοήθεια προς την Ελλάδα ε, εκταμιεύεται κατόπιν αιτήματος ε, της ε, ύπατος αρμοστίας ή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Διαπιστώνονται λοιπόν οι ανάγκες και εξετάζουμε πρώτα το εθνικό πρόγραμμα, κατόπιν εξετάζουμε τι απαιτείται τι πιστεύουν οι αρχές ότι χρειάζεται, αλλά και το τι πιστεύουν οι υπάλληλοι της Κομισιόν ε, στην ε, Κύπρο και την Ιταλία την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και άλλες χώρες ε, της πρώτης γραμμής. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, καθορίζουμε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα. Κάθε έργο όμως κατόπιν αξιολογείται με βάση τα, τη δική του αξία και τις ανάγκες. Ένα ε, παράδειγμα στην Ελλάδα είναι η στέγαση των ε, των προσφύγων, ε, διότι είναι πολύ ασταθής η κατάσταση. Έχουμε λοιπόν κάποιους καταβλισμούς, αλλά γίνεται συμπλήρωση με σκηνές ή με ξενοδοχεία αλλά προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε την πιο οικονομική λύση που να σέβεται όμως την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων. Όσον αφορά την Ιταλία, γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος Ιούνκερ κατέβαλε προσπάθειες να στηρίξει την Ιταλία στην κρίση μετανάστευσης. Ε, υποσχέθηκε επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τη χώρα και έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με τα Υπουργεία της χώρας ε, για να έχουμε ε, καλά προγράμματα. Έχουμε λοιπόν προγράμματα εκπαίδευση των ασυνόδευτων ανηλίκων, ε, προγράμματα για την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο και ασχολούμαστε και με την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης, της υπερεκμετάλλευσης των εργαζομένων. Κάποια από τα προγράμματα αυτά βρίσκονται ακόμα στη φάση του σχεδιασμού. Ελπίζω να απάντησε επαρκώ στι ερωτήσει σα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βιώτη. Ακόμα ένα ερώτημα. Για να καταλάβω. Δύο μάλιστα ερωτήσει. Να καταλάβω καλύτερα. Το πρώτο ερώτημα είναι να καταλάβω λίγο τη λογική που χρησιμοποιείτε. Γιατί η Ισπανία παίρνει τόσο λιγότερα λεφτά από την Ιταλία, μια και οι ροές ε, αυξήθηκαν στην Ισπανία σε σχέση με την Ιταλία. Ο, ο Ιταλός υπουργό Εσωτερικών λέει ότι στη χώρα μας μειώθηκαν ε, κατά 95% οι μεταναστευτικές ροές, ενώ αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές στην Ισπανία. Επομένως, τα νούμερα είναι τελείως διαφορετικά. Δεύτερον, η Κομισιόν συμφωνεί μαζί μας ε, μάλλον μπορεί να μας ενημερώσει για τα οικονομικά ε, σχέδια των κρατών μελών για το θέμα αυτό. Κομισιόν έχετε το λόγο. Το σχέδιο χρηματοδότησης υπάρχει για την Ελλάδα. Είναι ένα έγγραφο, μάλιστα, το οποίο είναι δημόσιο. Για την Ιταλία και για την Ισπανία έχουμε χρηματοδοτικά δελτία. Μπορούμε να σας τα δείξουμε. Ε, υπάρχουν και στην ιστοσελίδα μα κάποια από αυτά. Έχει, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τι ανάγκε που έχουμε εντοπίσει. Η Ιταλία, όπω σα είπα, ε, υπάρχει υπόσχεση του Ιούνκερ να υποστηρίξει την Ιταλική κυβέρνηση με 100 εκατομμύρια ε, πέρα ε, από αυτά που προβλέπονται στο εθνικό πρόγραμμα και εργαζόμαστε για αυτό το project εδώ και ένα χρόνο ε, τουλάχιστον, ε, γιατί θέλουμε να είναι καλά τα project. Αυτά δηλαδή ε, δεν αφορούν την πρώτη γραμμή υποδοχής, γιατί τα νούμερα εκεί έχουν μειωθεί πραγματικά πολύ στην Ιταλία, αλλά αφορούν την ένταξη των ε, ανθρώπων που είναι ήδη Για τους μετανάστες δηλαδή που έχουν λάβει το καθεστώς του δικαιούχου και μέτρα ε, εκπαίδευσης ασυνόδευτων ανηλίκων, ε, ανήλικοι που είναι ήδη στην Ιταλία. Η Ιταλία έχει πολλούς τέτοιους ανήλικους δικαιούχους, εν πάση και αιτούντες άσυλο. Για την Ισπανία είχαμε έντονο διάλογο με το Ισπανικό Υπουργείο και έχουμε εντοπίσει τις ανάγκες. Δεν μπορώ να σας πω τώρα στην αρχή της χρονιάς εάν ε, θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες με αυτά τα λεφτά, αλλά σε αυτή τη φάση αυτά χρειαζόταν η Ισπανική κυβέρνηση πέρα από αυτά που προβλεπόταν στο εθνικό πρόγραμμα. Το εθνικό πρόγραμμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ τα προηγούμενα χρόνια όπως στην Ιταλία ή στην Ελλάδα λόγω του χαμηλότερου αριθμού αφήξεων στην Ισπανία. Μέχρι τώρα όμως. Φυσικά αυτά αλλάζουν. Είναι πολύ ασταθής η κατάσταση. Ε, ακριβώς ε, αυτή είναι και η λογική της ε, βοήθειας αυτής. Προβλέπουμε επιπλέον χρηματοδότηση σε περίπτωση που χρειάζεται. Εστιάζουμε δηλαδή στις ανάγκες της, α, τη, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και ε, σας ζητήσαμε να συμφωνήσετε με αυτή τη μεταφορά. Εσείς και το Συμβούλιο ε, έχετε προτείνει 60 ε, εκατομμύρια στο αποθεματικό για το άσυλο. δεν έχουμε αποδεσμεύσει το ποσό, μπορεί να επανέλθουμε για επιπλέον λεφτά εάν χρειαστεί. Ευχαριστώ. Ο Γενικός Συγητής, παρακαλώ. Μία ερώτηση. Και για την Ιταλία. Μήπως ε, τα νούμερα τα οποία συζητάμε δεν έρχονται σε αντίθεση με την, Ιταλική, με την πολιτική της Ιταλικής κυβέρνησης που κλείνει τα κέντρα ε, για τους πρόσφυγες κτλ. Εγώ είμαι Ιταλό και σας τα λέω αυτά. Στι ε, περιφέρειές μα και στι κοινότητες και δήμους δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα για τα οποία λαμβάνουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου, πρέπει να μου απαντήσετε τώρα αμέσω, γιατί έχω πολλέ άλλε ερωτήσει. Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στι πολιτικέ τη Ιταλική κυβέρνηση που δεν παρέχει πια αυτέ τι υπηρεσίε και τη χρηματοδότηση που θέλουμε να δώσουμε στην Ιταλία. Μήπω υπάρχει αυτή έτσι, η σύγκρουση, η αντίφαση. Ε, κύριε Γενική η αν έχετε και άλλε ερωτήσει, να τι θέσετε τώρα, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο σε λίγο. Θα μα τελειώσει ο χρόνο. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι περίπλοκο όμω το θέμα. Εντάξει, να θέσω και τι άλλες ερωτήσεις. Μπορούμε και να το αναβάλουμε, έτσι. Μπορούμε να το αναβάλουμε. Εάν θέλετε επιπλέον διευκρινήσει. Δεν είμαστε αρκετά έτοιμοι ίσω. Εγώ έχω προτείνει να αναβάλουμε την ψηφοφορία γιατί υπάρχει πρόβλημα. Εφόσον προτείνετε αναβολή της ψηφοφορίας, εάν δεν έχετε μεγάλο πρόβλημα κομισιών, τότε καλό είναι να λάβετε αυτέ τι ενδείξει που θέλετε μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. αυτέ τι διευκρινήσει και τι εξηγήσει. Είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε για το 1 και το 7, για τα σημεία 1 και 7 και ζητάμε την αναβολή του 5 και του 8. Σωστό. Όμω, υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θέλω να θέσω. Πότε θα τα συζητήσουμε αυτά. Να τα, κάνουμε, να τα ρυθμίσουμε γραπτός. Πολύ γρήγορα, αν θέλετε τώρα. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα, λέει ο κύριο Βιώτη. Το θέμα είναι κάπω να επικοινωνήσω εγώ με την Επιτροπή. Και με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, Ελευθέρων ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να τα ρυθμίσουμε και γραπτό. Ακόμα καλύτερα, μάλιστα. Έτσι. Είναι ακόμα καλύτερα. Να μια λύση, λέει ο πρόεδρο. Γραπτό. Θα ψηφοφορήσουμε λοιπόν την α, μεταφορά 5. Ή μάλλον διορθώνει ο πρόεδρο. Θα ψηφίσουμε την 1 και την 7 τώρα. Έτσι. Ψηφίζουμε με ηλεκτρονική ψήφο τώρα. Ο κύριος Σολέ έχει μια ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την πρώτη πρόταση σχετικά με τη Συμφωνία Αλληλείας με το Μαρόκο, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για παράνομη συμφωνία, η οποία αντίκειται στη συμφωνία του δικαστηρίου διότι η Δυτική Σαχάρα δεν είναι έδαφος του Μαρόκου. Και γι' αυτό θα καταψηφίσω την πρόταση. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία, το καταγράφω αυτό, αυτή τη δήλωσή σας. Λοιπόν, για τη μεταφορά 1, υπαριθμών 1, ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας προφορίας, 10 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, καμία, μία αποχή. Και προστάθουμε και μία άλλη προφορική ψήφο, 11 ψήφοι υπέρ, για την ε, μεταφορά υπαριθμών 7. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας προφορίας. 12 συν 1, 13 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Ο Πολ Ρουμπίκ. Για τα άλλα τμήματα του προπολογισμού. Έχει το λόγο. Äh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τρεις τομείς όπου έχουν προταθεί ε, μεταφορές από το Κοινοβούλιο ε, και το Ελεγκτικό Δικαστήριο. Ε, έχουμε το C1 από το Κοινοβούλιο, έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό. 4,2 ε, εκατομμύρια στην ε, γραμμή 1400. Έχουμε να κάνουμε με τους 51 συμβασιούχους. Έτσι λοιπόν θα δημιουργηθούν 51 νέες ε, θέσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Η σύμβασή τους λίγη 31 Ιουλίου και προτείνεται να συνεχίσει η απασχόλησή τους από την Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ, το Κοινοβούλιο. Θέλει να παρατείνει τις συμβάσεις τους μέχρι το 2019. Σας ευχαριστώ πολύ. Για αυτό το σχέδιο μεταφοράς τώρα. Ποιος θέλει το λόγο, ο κύριος Ντεπρέ. Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση για την προέλευση των κονδυλίων που μεταφέρονται. Όλοι συμφωνούμε για το ότι η ασφάλεια των κτηρίων και η γενική ασφάλεια, έτσι είτε του κυβερνοχώρου είτε των κτηρίων, είναι προτεραιότητα για μας. Και έχουμε φροντίσει να υπάρχουν τα αναγκαία κονδύλια. Διαπιστώνω όμως ότι εδώ θα αποσύρουμε 127.000 ε, ευρώ, τα οποία καταρχήν θα πηγαίνανε στη γενική ασφάλεια των νέων ε, κτηρίων και τα παίρνουμε από εκεί και τα βάζουμε στην ε, παράταση της σύμβασης των 51. Δεν με έπεισε η απάντηση που άκουσα πριν. Εγώ δεν πίστηκα για την αναγκαιότητα της παράτασης της σύμβασης των 51 αυτών. Οπότε, αφού έχουμε τονίσει τόσο πολύ την ασφάλεια και των κτηρίων και του κυβερνοχώρου, για μένα δεν είναι αναγκαία η παράταση αυτή. Οπότε θα ήθελα να μου το εξηγήσετε αυτό. Προέδρο, θα μας απαντήσουν βέβαια μετά από την Επιτροπή, η κυρία Καζιαβδάλ. Ευχαριστώ. Παίρνω το λόγο για να επανέλθω σε μία ερώτηση που έκανα και νωρίτερα, γιατί δεν είναι για μένα ξεκάθαρο. Τα χρήματα, τέλος πάντων το τιμήμα. με διαφορά με τον κύριο ε, Ντεπρέ, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα να διατηρηθούν οι συμβάσει των 51, γιατί καταλαβαίνω ότι το έργο τους έχει κάποιες θετικές επιπτώσεις, αλλά δημοσιονομικά εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω πώς αιτιολογούνται 3,3 εκατομμύρια ευρώ για 5 μήνες, για 51 άτομα. Εξακολουθώ να μην το καταλαβαίνω. Και δεύτερον, αν μπορεί κάποιο να μου απαντήσει τώρα έχει καλός, αλλιώς να μας απαντήσουν όταν μπορούν, το στομότερο δυνατόν. Αλλά πιστεύω ότι αφού μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο συνδέεται άμεσα με τον προπολογισμό το 2020 και θα ήταν ε, παράλογο να αποφασίσουμε τώρα για τους πέντε μήνες χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει το 2020, θα ήταν λογικό να καθυστερήσουμε αυτή την ψηφοφορία, να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα που θα γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Προεδρείο. Αλλά από τις δικές μου τις πληροφορίες, τα 3,3 εκατομμύρια για 5 μήνες, για 51 ανθρώπους, δεν μου βγαίνει εμένα αυτός ο λογαριασμός. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάς τώρα να απαντήσει. Τι γίνεται με την ασφάλεια των κτηρίων, πλήτεται. Για το θέμα της ε, ασφάλειας, ναι, γιατί για το άλλο δηλαδή την ανάλυση των ποσών. Είναι ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας που μπορεί να απαντήσει. Αλλά για την ασφάλεια, με δύο λόγια πρόκειται για την φύλαξη των κτηρίων Αντενάουερ στο Λουξεμβούργο, όπου υπήρξε μια καθυστέρηση και προσαρμόστηκε τώρα το χρονοδιάγραμμα πιο ρεαλιστικά. Οπότε το κτίριο έτσι κι ε, δεν θα έχει το προσωπικό του το 2019, αλλά αρχές του 2020. Οπότε δεν χρειάζεται να υπάρξει μια φύλαξη όπως είχαμε προβλέψει. Για την ανάλυση τώρα των ποσών στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, είναι εδώ κυρία Ρούτε, στη διάθεσή σας για να σας απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Παρακαλώ, εσείς. Για αναλύστε μας τα ποσά, πώς εξηγούνται. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, πανέλθω λίγο σε αυτά τα ποσά. Πράγματι, ζητήσαμε 4 εκατομμύρια το 2018. Η πρόληψη ξεκίνησε όταν έγινε μεταφορά δηλαδή ανάμεσα στο Μάρτιο και τον Ιούλιο. Εμείς προσλάβαμε ε, τους 51 ε, υπαλλήλου και άρχισαν να δουλεύουν αλλά με διαφορετική ημερομηνία ο καθένας. Οπότε τώρα δεν πρόκειται μόνο για αυτούς τους 51, δεν είναι για 5 μήνες, η σύμβαση είναι μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Οπότε θέλουμε να προχωρήσουμε για 5 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο και θέλουμε επίσης να παρατείνουμε και κάποια διαρθρωτική ενίσχυση. Για παράδειγμα, πολύ ειδικευμένου που δεν έχουμε στο προσωπικό μας. Δημιουργείται, για παράδειγμα, μία μονάδα ε, σύλληψης και σχεδιασμού. Είπαμε ότι αυτή τη φορά δεν θα πάμε σε εξωτερικούς υπαλλήλους, για την εκστρατεία μας ε, προκειμένου να πάνε οι πολίτες να ψηφίσουν, αλλά θέλουμε μία μονάδα που θα φωσιωθεί αποκλειστικά ε, στο να μας προσφέρει υλικό που συνήθως μας δίνουν εξωτερικοί. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε designers, ειδικού στο copyright, που δεν έχουμε στο προσωπικό μας. Οπότε τα 3,3 εκατομμύρια για τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας καλύπτει τις συμβάσει για τους 51, αλλά και την ενίσχυση επίσης στα κέντρα μας στις Βρυξέλλες. Και όλα αυτά εξηγούνται στις πληροφορίες για τη μεταφορά που έχετε στη σελίδα 2. Πρόεδρος, ωραία. Ε, αναβολή ζήτησε κάποιος. Κύριε και εσείς τι λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με το ότι το Κοινοβούλιο ασχολείται περισσότερο με την επικοινωνία και ότι θέλει να γίνεται πιο επαγγελματικά η δουλειά αυτή. Νομίζω ότι υπό το φως της συνδιαλλαγής είναι σωστό να συζητήσουμε πώς θα προχωρήσει το θέμα. Εμένα λοιπόν θα με ενδιέφερε τι μορφή θα έχει η δουλειά αυτή το 2020 και αν υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει. Ο εισηγητή μα, ο κύριο Μάνκα, μα είπε ότι πρότεινε να διατηρηθούν αυτέ οι 51 θέσει στον προπολισμό του 2020. Ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι όχι μόνο γιατί, κοιτάξτε, υπάρχουν τα άτομα αυτά που τα χρειαζόμαστε και εξάλλου πρόκειται για ενίσχυση της προβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε εμείς μέχρι το τέλος παρατείνουμε τις θέσεις αυτές. Αυτό θέλουμε αλλά πράγματι αυτό εξηγείται γιατί τα άτομα αυτά προσφέρουν σημαντικό έργο. Θα έπρεπε να συνεχίσουν με το έργο τους. Αποτελούν προστιθέμενη αξία για μας. Και γι' αυτό θέλουμε να υιοθετήσουμε αυτή την απόφαση. Να διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε δηλαδή αυτούς τους 51 αλλά νομίζω ότι έχει υποθεί ξεκάθαρα από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία ότι του χρειάζονται αυτού του ανθρώπου. Και εγώ το στηρίζω για το 2020, ναι. Ευχαριστώ. Κύριε Ρούμπικ, τι θα κάνουμε, θα ψηφίσουμε τώρα ή αναβάλλετε η ψηφοφορία. Τι μας λέτε. Θα ήθελα ε, να ακούσω την θέση της Κομισιόν. Πώς βλέπουν το έτος 2020 και πιστεύει ότι ε, αυτοί οι 51 συμβασιούχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται και το 2020. Σύντομα παρακαλώ απαντήστε μας. Πολύ σύντομη δεν ε, μετράμε τις ε, θέσεις ε, στο σχέδιο μας. Εξετάσαμε τα προφίλ των συμβασιούχων και θα συνεχίσουμε να τους θεωρούμε συμβασιούχους στα γραφεία μας. Δεν έχουμε σχεδιάσει λοιπόν τη δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων. Oui, mais vient un moment où le... Ναι, αλλά η παράταση των συμβάσεων δημιουργεί υποχρεώσεις. Αν διακοπεί η σύμβαση μετά. Ωραία, λοιπόν, θα ψηφίσουμε τώρα ή τη Δευτέρα το βράδυ. Η πρότασή μου είναι πρώτα να ε, κάνουμε τη συνδιαλλαγή και να ψηφίσουμε την επόμενη φορά. Ωραία, ψηφίσουμε Δευτέρα βράδυ. Για τα άλλα αιτήματα μεταφοράς, κύριε Σιγητά, θα είναι πιο εύκολο, έτσι δεν είναι. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να εργαστούμε γρήγορα. Ε, Ε, το C2 είναι 64.000 ευρώ για την ε, μεταφορά δεμάτων. Έχουμε αλλάξει συνεργάτη. Ε, προτείνω να υιοθετήσουμε την πρόταση. Πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Επιτροπή Περιφερειών. Και όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών, ε, έχουμε τροποποίηση όσον αφορά το προσωπικό, δύο μόνιμες θέσεις της κατηγορίας 4. και η μόνιμη θέση γραμματέα και μία θέση γραμματέα στην ε, κατηγορία 5 θα πρέπει να γίνουν προσωρινές θέσεις. Συμφωνώ, διότι ουσιαστικά πρόκειται απλά για μετατροπή των ε, υπάρχουσων θέσεων. Τρία αιτήματα για μεταφορές έχουμε για το ελεγκτικό συνέδριο. Ναι, έχουμε τρεις ε, γραμμές... Ε, έχουμε τρεις γραμμές για το ελεγκτικό συνέδριο. Έχει να κάνει με συμβασιούχους. Ε, μιλάμε για αύξηση και για τα σχετικά συστήματα πληροφορικής, για τη συντήρησή τους. Η δεύτερη γραμμή είναι καθαρισμός και συντήρηση, όπου επίσης προβλέπεται ε, αύξηση για την ηλεκτρική θέρμανση και τον κλιματισμό, καθώς και μια μετατροπή ε, θέσης βοηθού από την κατηγορία 3 στην κατηγορία 5 και ε, την υπηρεσία δημοσιεύσεων. Ε, είμαι υπέρ. Πολύ ωραία. Η επόμενη μεταφορά. Όχι, αυτά είναι όλα. Ωραία. Για τα πέντε τίματα αυτά, για μεταφορές κονδυλίων. Υπάρχουν ερωτήσεις μήπως? Σουατ, όχι. Αν δεν υπάρχουν ούτε ερωτήσει ούτε αντιρρήσει, εγκρίνονται αυτέ οι αιτήσει μεταφορά. Έτσι. Ωραία, εγκρίνονται. Και τώρα, η Μόνικα Χολμέγερ έχει το λόγο για να μας μιλήσει για την υπηρεσία φαρμάκων, το κτίριο της υπηρεσίας φαρμάκων. Ah, Α, ah, όχι, ο κύριος Ντεπρέ θα μας τα πει. Αντικαθιστά την κυρία Χολμέγερ. Εντυπωσιακό, πρόεδρε. Γιατί, λέει ο πρόεδρος. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ήδη συζητήσει στην τελευταία μας συνεδρίαση. Ο Οργανισμός Φαρμάκων. Όσοι ξέρουν το φάκελο, ξέρουν περί πρόκειται ε, είναι κατεστημένος οργανισμός στο Λονδίνο, στο μεταξύ έγινε το Brexit. Επομένως, ο οργανισμός φαρμάκων δεν χρειάζεται τα κτίρια αυτά που νίκιασε. Δυστυχώς, όμως, δεν έχει ρήτρα λύσης του συμβολέου στην σύμβαση που υπογράφτηκε. Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει το νίκη σε περίπτωση που δεν μπορούσε να υπενικιάσει ε, τα κτίρια αυτά, να βρει κάποιον που θα δεχόταν να τα υπενικιάσει, εν όμως ο ιδιοκτήτης δεν είναι σίγουρος ότι θα πληρωθεί το νίκη ε, από εδώ και πέρα. Θέλει επιπλέον λοιπόν εγγύησεις. Ποια είναι τα τεχνικά στοιχεία λοιπόν του φακέλου. Σας διαβάζω αυτά που μου γράφει η κυρία Χολμάιερ. Ζητάτε από την Δημοσιονομική Αρχή να εγκρίνει μία ε, επιχείρηση για τα κίνητα που θα έχει επίπτωση, ε, γιατί θα φτάσει μέχρι τα 67 εκατομμύρια, ε, εκατομμύρια. Τα 36 εκατομμύρια θα πρέπει να χρηματοθούν, τα 28 υπόλοιπα έχουν καταβληθεί με βάση την αποδε... αποδεδειγμένη δημοσιονομική τεχνική. Ε, πρώτο σημείο. Μπορούμε να φτάσουμε 67 εκατομμύρια και αφορά τα 38,7 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό που μένει, δύο. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι η Κομισιόν κάνει το κατά για να υποστηρίξει τον ΕΟΦ στον, στη διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη. Πιο συγκεκριμένα, η συγκήτρια καλεί την Κομισιόν να κάνει το κατά δύναμη ώστε να δώσει τις απαραίτητες εγγύσεις στον ιδιοκτήτη μέσω μίας επιστολής, ούτω ώστε ο ΕΟΦ να μπορέσει να συνάψει αυτή τη συμφωνία ε, με ικανοποιητικέ συνθήκες το συντομότερο δυνατόν. Ο, η εισηγήτρια ζητάει επίσης η Κομισιόν να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ΕΟΦ και τον ιδιοκτήτη, γιατί αυτό θα ενισχύσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις απέναντι στον ιδιοκτήτη. Η εισηγήτρια θεωρεί επίσης ότι οποιοδήποτε μετοντικό κόστος για τον ΕΟΦ που απορρέει από, μη, από αδυναμία πληρωμής ε, του, της επιρρενικίασης θα πρέπει να προέλθει όχι από το κονδύλι του ΕΟΦ, αλλά από τον προπολογισμό της Ένωσης. Τέλος, θα πρέπει να δοθούν αρκετά κονδύλια σε περίπτωση στην, στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για να καλύψουμε όλο το επιπλέον κόστος που θα προκύψει για τον ΕΟΦ λόγω της υποχρέωσης που έχει να τιμήσει τη σύμβαση ενοικίαση στο Λονδίνο. Κάνει και κάποιες συστάσεις, θα σας διαβάσω. Συστήνουμε λοιπόν να εγκρίνουμε τη σύμβαση και τις οικονομικές επιπτώσεις που σας έχω απαριθμίσει. Μιλάμε για 38,7 εκατομμύρια, έτσι που υπολείπονται. 38,7 εκατομμύρια ευρώ εκεί ευρώ. Και να γράψουμε το εξή στα πρακτικά. Η Κομισιόν θα πρέπει να υποστηρίξει τον ΕΟΦ στι διαπραγματεύσει με την ε, ομάδα Κάντρου Γουόρφ και να ε, μιλήσει με την ε, Βρετανική κυβέρνηση. Καλείται επίση η Κομισιόν να κάνει το με το σώστο να δώσει τι απαραίτητε εγγυήσει στον ιδιοκτήτη. Ε, μιλάει για την περίπτωση που πρέπει να σταλεί μία επιστολή, ούτω ώστε ο ΕΟΦ να μπορέσει να συνάψει αυτή τη σύμβαση. Επίσης, ε, υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, να και ένα καλό νέο, είχε εκφράσει σημαντικές επιφυλάξεις το 2011 σε ό,τι αφορά την υπογραφή μιας σύμβασης ενοικίαση χωρίς ρήτρα λύσης της σύμβασης αυτής. Επίσης, υπενθυμίζει ότι το κόστος για τον ΕΟΦ αποφασίζει από την απόφαση των κρατών μελών και επομένω το Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει του απαραίτητου πόρου για να αντιμετωπίσει ο ΕΟΦ τις συνέπειε αυτή τη απόφαση. Αυτά, Πρόεδρε, νομίζω ότι θα έπρεπε να δώσουμε το λόγο στον Οργανισμό Φαρμάκων για να μας επιβεβαιώσει ε, αυτά τα στοιχεία ή να μας δώσει περισσότερες ε, πληροφορίες για όλα αυτά και συνεχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς αντιδρά ε, απέναντι σε αυτά τα αιτήματα της εισηγήτριας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ποιος εκπροσωπεί εδώ τον Οργανισμό Φαρμάκων? Παρακαλώ. Θα κούνες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ για τα όσα είπατε. Πράγματι, στο στάδιο αυτό θέλω να αναφέρω ότι δεδομένου ότι δεν έχουμε να προτείνουμε ποινικίαση, η συναλλαγή αυτή θα ήταν προς όφελος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου και των, του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Και όντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα θέλαμε να συμφωνήσει με την πρόταση αυτή και για τα κονδύλια τα οποία αναφέρονται στην πρόταση. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστως να σας απαντήσουμε. Πρόεδρος. Δεν έχετε ιδιαίτερε παρατηρήσεις για το όσο είπε ο κύριος Ντεπρέ. Σας φαίνονται καλά και σύμφωνα με τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου για αυτή την περίπτωση, έτσι, συμφωνείτε δηλαδή. Ωραία, Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών. Τι λέει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεπρέ που συνόψιζε τη θέση της εισηγητρίας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τον οργανισμό στη διαπραγμάτευση αυτή. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο αντίκτυπος του 67% ε, ε, θα ε, γίνει αισθητό μέσω ή αμέσω στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δεν προτείνει κανείς τροποποίηση στην δομή του προϋπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτηθεί αυτό από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφέ ότι το 2019 αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του ισχύοντο προπολογισμού και τη επιχορήγηση ε, του οργανισμού. Για το έτος 2020 όμω είναι σαφέ ότι στο σχέδιο προπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει υψηλότερη επιχορήγηση ε, που θα ήταν ε, αυτό που θα ίσχυε κανονικά και που ίσχυε τα προηγούμενα έτη. Το άλλο σημαντικό στοιχείο που ανέφερε ο κύριος Ντεπρέ είναι το θέμα της επιστολής και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο ε, Επίτροπος Έτιγκερ σκοπεύει να στείλει τέτοια ε, επιστολή ε, στον ε, εκμιστοτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τον οργανισμό και θα τις παράσχει τους απαραίτητους πόρους για να τηρήσει τις ε, συμβατικές της υποχρεώσεις ε, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με την υπενικίαση. Και ελπίζουμε ότι με μια τέτοια καθησυχιαστική επιστολή προς τον εκμισθωτή, ο οργανισμός θα μπορέσει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τον υπενικιαστή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντεπρέ, ακούσατε δύο παρεμβάσεις που είναι προς την κατεύθυνση των συστάσεων που εσείς μας αναφέρατε εκ μέρους της κυρίας Χολμάγερ. Ναι, Πρόεδρε, όντως σημειώνω την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την επιστολή, αλλά θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος για τα ποσά. Οπότε γι' αυτό ρωτάω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκατε σε 27 εκατομμύρια, αλλά εγώ ξέρω ότι 28,2 από αυτά έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί. Άρα παραμένει ένα ποσό 38,7 προσκάλυψη. Απάντηση. Ναι, ορθά. Το πρώτο τμήμα χρηματοδοτείται ήδη το 2019 και το υπόλοιπο το 2020. Δεν πρέχω και άλλη μια ερώτηση. Γιατί στις συμβάσεις αυτού του τύπου υπάρχουν πάντα ρήτρε προσαρμογής του ενοικίου. Μήπω κινδυνεύουμε να έχουμε κάποια κακή έκπληξη, δηλαδή ο ιδιοκτήτης έτσι, για την προσαρμογή της μίσθωσης. Μήπως μέχρι το τέλος της περίοδου που καλύπτει η σύμβαση θα έχουμε μια άσχημη έκπληξη γιατί θα μας πει ο ιδιοκτήτης ότι αποφάσισε να αυξήσει την τιμή του ενοικίου. και το μίστομα να αυξηθεί. Πρόεδρος, δηλαδή αν αυτός που επινοικιάζει δεν πληρώσει, θα έπρεπε να πληρωθεί το ποσό από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, σωστά. Αυτό θέλουμε να προβλέψουμε. Εξού και η επιστολή. Δηλαδή, είμαστε στο έλεος το διοκτήτη. Δηλαδή βασικά αν κάτι δεν πάει καλά την πατήσαμε. Δηλαδή αναλαμβάνουμε μια δέσμευση, εντάξει όχι για 67 εκατομμύρια, αλλά για 500. Γιατί αν αύριο μεθαύριο, εντάξει μπορεί να υπερβάλλω στο νούμερο, αλλά θέλω να πω ότι αν αυτός που επινοικιάζει δεν πληρώνει, αν δεν βρούμε άλλον, θα πρέπει να πληρώσουμε. όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ε, αυτό το επιπλέον ε, άνοιγμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 67 εκατομμύρια. Η σύμβαση του οργανισμού και με το σενάριο της υπενικίασης θα πρέπει να επανεξετάζεται κάθε πέντε χρόνια ε, το ενίκιο ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς, αλλά εφόσον θα πληρώνεται από υπενικιαστή, εάν υπάρξουν ε, αντίστροφες ε, τάσεις, δεν θα είναι υποχρεωμένος ο οργανισμός να πληρώσει. Ο υπενικιαστής λοιπόν, θα πληρώσει τη διαφορά κατευθείαν στον εκμισθωτή. Μετά, λοιπόν, από την συναλλαγή αυτή, δεν θα πρέπει να υπάρχει άνοιγμα πια για τον οργανισμό για τη σύμβαση αυτή που θα ισχύει μέχρι το 2039, για 20 χρόνια δηλαδή. Όσον αφορά τις εγγυήσεις, ε, οι κίνδυνοι θα υπάρξουν, κίνδυνοι αθέτησης στο μέλλον. Ε, ελπίζουμε αυτό να μην συμβεί. Θεωρητικά όμως υπάρχει ο κίνδυνος. Ο οργανισμός στις διαπραγματεύσεις ε, κατάφερε να λάβει εγγύηση από την γονική εταιρεία, τη μητρική εταιρεία, η οποία θα καλύψει ε, τα ε, κίνητρα αυτά προς ε, τον υπενικιαστή. Θα υπάρξει δηλαδή εγγύηση από πλευράς της μητρικής εταιρείας. Δηλαδή θα παρέμβει ο οργανισμός φαρμάκων. Σε περίπτωση αφέτησης από τον υπενικιαστή, η γονική εταιρεία θα παρέμβει και θα υπάρξει ένα διάστημα χωρίς εγγύηση για τον οργανισμό, το διάστημα δηλαδή που θα αναζητείται άλλος υπενικιαστής. Και, Όταν μιλάτε για άλλο οργανισμό, τι εννοείτε. Εννοώ ότι έχουμε μητρική εταιρεία, αμερικανική. Μητρική εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την υπενικίαση και θα υπάρξει ένα μέσο ειδικού σκοπού για την υπενικίαση των εγκαταστάσεων. Ναι, ναι. Άμα καταλάβατε, σας φαίνεται ξεκάθαρο. Ο κύριος Ντεπρέ. Πρόεδρε, εγώ απλώς μετέφερα τα λόγια της κυρίας Ολμαγερ. Κίνη ζητάει η αρχή επί του προπολογισμού να εγκρίνει την, το ποσό που πρέπει να καλυφθεί για αυτή τη συναλλαγή την κτηριακή, το σύνολο των 67 και μένει το 38,7 πρέπει να καλύψουμε. Και η Επιτροπή πρέπει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον οργανισμό και τον ιδιοκτήτη για να ενισχυθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε ε, κόστος το οποίο θα προκύψει από τον επινοικιαστή θα πρέπει να πληρωθεί από τον προπολογισμό της Ένωσης. Αυτή είναι η απόφαση εκ μέρους της κυρίας Χολμάγερ που ζητάω να εγκρίνει η Επιτροπή μας σήμερα. Πρόεδρος, ωραία, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. 10 υπέρ. 11. 11 υπέρ. Η κυρία Ολμάγερ ευχαριστεί την Επιτροπή μας, λέει ο κύριος Δεπρέ. Πρόεδρος, ε, η Επιτροπή μας ευχαριστεί την κυρία Ολμάγερ. Τώρα, τι άλλο έχουμε. Θα ακούγαμε την κυρία Ολμάγερ και όσον αφορά κάποια σχέδια για κτίρια που δεν χρησιμοποιούμε των οποίων είμαστε όμως ενοικιαστές ή ιδιοκτήτες, αλλά αυτό το σημείο να βάλετε για την επόμενη εβδομάδα. Διάφορα. Ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα και θα μιλήσω πορτογαλικά. Από την προηγούμενη εβδομάδα ένας κυκλώνας έπληξε το Μαλάου, τη Μοζαμβίκη και οι επιπτώσεις ήταν καταστροφικές, ιδίως στον Πίρακ 70% των εγκαταστάσεων καταστράφηκαν, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό. Υπάρχουν πάνω από χίλιοι νεκροί και πάνω από 100.000 έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κατάσταση είναι πολύ έκτακτη, όπως καταλαβαίνετε, και θα έπρεπε να διαθέσουμε όλα τα μέσα που μπορούμε. Είναι σημαντικό το μήνυμα αυτό να περάσει στον κύριο Γιούνκερ και στον κύριο Στυλιανίδη επίσης. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Σας στηρίζουμε. Έτσι. Κύριε Ντεπρέ, έχετε εντολή για να μας παρουσιάσετε και τις πληροφορίες για τα κτίρια και τις υποδομές. ναι, να ψάξω να βρω το έγγραφό μου. Πρόκειται για ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας ενημερώνει για τα εξής. Ανάμεσα στο 2019, τώρα δηλαδή, και το 2025, η ενοικίαση για 165.000 τετραγωνικά μέτρα που καλύπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες εκπνέει ανάμεσα στο 2019 και το 2025, 165.000 τετραγωνικά μέτρα. Όμως, και εδώ ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει, όσον αφορά τα έτη 2020-2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει με προσφορές και ψάχνει κτίρια για να έχει στη διάθεσή τη 80 με 150.000 τετραγωνικά μέτρα. Οπότε ελευθερώνονται 165.000 τετραγωνικά μέτρα, αλλά ανάμεσα στο 2020 και το 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψάχνει να νοικιάσει 80.000 με 150.000 τετραγωνικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως θα μπορούσε να μας το εξηγήσει αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στην ψαλίδα των ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας εξηγήσει ή τέτοια ώρα να το αφήσουμε για την επόμενη συνεδρίαση. Απάντηση. Ναι, και εγώ ψάχνω εδώ πέρα πεγνωσμένο, αλλά δεν βλέπω και τους συναδέρφους, οπότε ναι, να σας απαντήσουμε γραπτά, παρακαλώ. Πρόεδρος μπορούμε να το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη μια επόμενη συνεδρία τη επιτροπή μας. Ωραία, δεν έχει ζητήσει κανεί το λόγο. Ωραία, επόμενη συνεδρίαση είναι 25 Μαρτίου, σε μία εβδομάδα δηλαδή, στις 8 το βράδυ στο Στρασβούργο. Και 1η και 2 Απριλίου εδώ στις Βρυξέλλες πάλι. Κυρίσω τη λήξη τη συνεδρίασης.